ύμνο που θα ερμηνεύσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Στρασβούργου, το Ρέμι Άμπραχαμ. Ευχαριστούμε τον Μαέστρο, ευχαριστούμε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη βάση του άρθρου 14 εδάφιο 2 του ιστορικού κανονισμού υπό την προεδρία του απερχόμενου Προέδρου δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία συζήτηση Ε, της οποίας το θέμα δεν σχετίζεται με τον έλεγχο της εντολής ή την ε, εκλογή των προέδρων.